Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Να ξεκινήσουμε αμέσως. Please take seat. Παρακαλώ, καθίστε. Καλημέρα σας. Ένα θερμό καλωσόρισμα στον προσκεκλημένο μας, τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντέισελμπλουμ, τον οποίο ευχαριστώ που ήρθε σήμερα εδώ, για να συμμετάσχει στον πρώτο γύρο οικονομικού διαλόγου για την νέα 8η θητεία του Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, ο οικονομικός διάλογος είναι ένα θεμελιώδες σκέλος της λογοδοσίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμενού και η σημερινή συζήτηση με τον κύριο Ντέισιμπλουμ μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τις αναχώρασεις τάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο από το Συμβούλιο. σημαίνοντας έτσι την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014. Θα μπορέσουμε όμως να συζητήσουμε και γενικότερα ζητήματα που μας απασχολούν για την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, τα εργαλεία διακυβέρνησης, το γνωστό θέμα για τις επενδύσεις, την ευελιξία και ούτω καθεξής. Είχαμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εχθές για το πώς οι αναχώραση τάσεις έχουν υλοποιηθεί ως τώρα και ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αποφεληθούμε από τη σημερινή επίσης συζήτηση ώστε να ε, προωθήσουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο. Βάσει των διατάξεων του νομικού πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να ελέγξουμε, να ελέγξουμε όλα τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όλα τα μέτρα που έχει λάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να θυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτός ο κύριος οικονομικού διαλόγου με τον πρόεδρο του Eurogroup προβλέπεται δίσετησίως. Και να σας θυμίσω και τη μέθοδο που ακολουθούμε συνήθως εδώ. Ο κύριος Τέισιμπλουμ θα κάνει την εισηγήσή του για 10-15 λεπτά και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν 5 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Εάν επίσης έχουμε χρόνο θα έχουμε και περαιτέρω συζήτηση. Θα παρακαλέσω θερμά τους συναδελφούς να μην εξαντλήσουν τα πέντε λεπτά τους για τις ερωτήσεις τους, διότι αν το ερώτημα τους διαρκεί τέσσερα λεπτά, ο συνομιλητής τους θα έχει ένα λεπτό για να απαντήσει μόλις. Παρακαλώ λοιπόν να διαχειριστείτε συνετά το χρόνο σας. Οι πολιτικέ ομάδε ήδη έχουν αποβάλει του αγορητέ του, οπότε δίνω ευθύ αμέσως το λόγο στον πρόεδρο του Eurogroup. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Με μεγάλη χαρά έρχομαι για μια ακόμη φορά ε, στην Επιτροπή σας, την πρώτη βέβαια μετά τις ευρωεκλογέ. Βλέπω κάποια γνωστά πρόσωπα αλλά και πολλά ε, καινούρια και περιμένω να ανταλλάξουμε απόψεις και να αποφελθώ και εγώ από την εμπειρία σας. Η έναρξη της νέας νομοθετικής περίοδου είναι μια καλή χρονική στιγμή για να κάνουμε έναν απολογισμό της οικονομικής κατάστασης και να θέσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωομάδας. Και αυτό θα πράξω υπό το πρίσμα των βασικών συστάσεων πολιτικής στον τομέα της Ευρωζώνης, τις οποίες εγκρίναμε τον Ιούνιο και τις οποίες δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε όπως λοιπόν ορίζεται και στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωομάδας, πρόθεσή μας είναι να συζητήσουμε την υλοποίηση των συστάσεων και την παρακολούθησή τους και αυτό θα γίνεται σε κάθε επόμενη συνεδρία της Ευρωομάδας. Αρχικά κάποια λόγια για την οικονομική κατάσταση. Τις τελευταίες, τις εβδομάδες ε, ο τύπος ε, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις εκτιμήσεις για τα δεδομένα του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, βάσει των οποίων το ΑΕΠ έχει παραμείνει σταθερό στην Ευρωζώνη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014 και έχει αυξηθεί κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2013. Τώρα, Αυτά τα βασικά ε, στοιχεία ε, ουσιαστικά κρύβουν ε, διαφορές ό,τι αφορά τις επιδόσεις. Έχουμε ισχυρότερες επιδόσεις σε χώρες όπως Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Οστανία, Σλοβακία, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται με τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποδίδουν, έχουν αποτελέσματα στις χώρες αυτές. Όμως ε, δεν είναι αρκετές αυτές οι ισχυρέ επιδόσεις για να αντισταθμίσουν απώλειες ε, και απώλεια αριθμού σε άλλες ε, χώρες και μάλιστα από τις μεγαλύτερες οικονομίες όπως η Γερμανία. Στη Γερμανία αυτή η απώλεια ο ρυθμού ίσως μπορεί να οφείλεται και σε μια πολύ, στις πολύ ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αλλά και σε ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις όπως η Ουκρανία και την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξελίξεις και όλα αυτά επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα ε, και το δημόσιο αίσθημα. Παραμένει πάντως ε, ε, εύθραυστη, παραμένουν εύθραυστα τα στοιχεία ανάκαμψης και δεν έχουμε ισορροπημένη ανάκαμψη σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν μπορώ να προκαταλάβω, θα γίνουν οι συζητήσει στο Μιλάνο την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των ε, Υπουργών Οικονομικών. Πάντω πρέπει να δώσουμε νέα όθηση ε, στι προσπάθειε μα για ανάκαμψη και μεταρρυθμίσεις. Παραμένουν οι ίδιε θεμελιώδει προκλήσει στην Ευρωζώνη και έχουμε θεσπίσει μια σαφή απάντηση πολιτική. Πρώτα απ' όλα στόχο μα είναι να μειώσουμε τα επίπεδα του δημόσιου και ιδιωτικού χρέου. Δεύτερον, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Και τρίτον, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να μπορέσει αυτός να λειτουργήσει προ όφελο τη πραγματική οικονομία. Κάτι που χρειαζόμαστε και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ώστε ε, να επανέλθουν ε, τα επίπεδα εκεί που ήταν ε, τα τελευταία χρόνια. Πριν την τελευταία δεκαετία που είχαμε συνέχεια επιδεινούμενα επίπεδα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ήδη στην Ευρωζώνη ήταν πολύ θαραλέα ε, και έχουν δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα βάσει στα οποία θα πρέπει να ε, χτίσουμε. Έχουμε κάνει πρόοδο για να επανέλθει σε μια βιώσιμη κατάσταση ο τομέας των δημοσίων οικονομικών. Προβλέπεται το μέσο έλλειμμα στην Ευρωζώνη κάτω από τα 3% του ΑΕΠ στο 2014 και υπάρχουν χώρες ε, ε, με υπερβολικά ελλείμματα μεν ε, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά μειώνεται ο αριθμό των χωρών αυτών. Η απομόχληση στον ιδιωτικό τομέα προοδεύει και έχουμε σταθερότητα στις αγορές ε, του δημόσιου χρέους και είχαμε και σημαντική μείωση στις αποδόσεις των ομολόγων σε πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να κάνουμε διπλές προσπάθειες για να δημιουργήσουμε μία ε, βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να βρούμε το σωστό μείγμα πολιτικής συνδυάζοντας τι προσπάθειές μας ώστε να έχουμε ε, φορολογικές πολιτικές ε, φιλικές προς την ανάπτυξη. να αντικατοπτριστούν ε, και στου εθνικού προπολογισμού, στα σχέδια των εθνικών προπολογισμών. Πρέπει να προωθηθούν αυτέ οι επιθρεπτικέ μεταρρυθμίσει ε, για να προωθηθεί και η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι κεντρικό στοιχείο τη στρατηγική μα για να βγούμε από την κρίση. Πολλέ μεταρρυθμίσει ήδη έχουν δρομολογηθεί για τι αγορέ εργασία, αγορέ προϊόντων, και μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να πω ότι ανάλογα με το κράτος μέλος ε, διαφορετικές ε, είναι οι κατάλληλες, ε, κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Το στόχος είναι όμως να μεγιστοποιήσουμε τα συλλογικά ωφέλη. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρωομάδας. Με όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν ε, το επόμενο εξάμεινο μια σειρά συζητήσεων για διαθροτικές πολιτικές. Ήδη αρχίσαμε να, να συζητούμε τα μέτρα και σχέδια των κρατών για να μειωθεί το υψηλό μη μισθολογικό κόστος εργασίας που πάντοτε αποτελεί ε, πρόκληση σχεδόν για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης ε, που έχουν ένα φορολογικό βάρος εργασίας υψηλότερο από το μεσόρο του ΩΣΑ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος και εμπόδιο για την ανάπτυξη. Ε, και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα εξετάσουμε λοιπόν μια δέσμη κοινών αρχών, βέλτιστων πρακτικών, ε, θα τα εξετάσουμε την επόμενη εβδομάδα, όπως επίσης ε, θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και τα σχέδια για μειώσεις του μη κόστους και άλλες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις το φθινόπωρο όταν θα συζητήσουμε τα σχέδια προπολισμού των κρατών μελών. Πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτήμου, στο peer review, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συντονισμό ε, δημοσιονομικό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και Βέβαια στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι συστάσεις αναχώρα ε, και αυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη του οι χώρες όταν θα καταρτίζουν το σχέδιο προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας ε, κατακαιρματισμός. Δεν θέλουμε ε, να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός και νομίζω ότι κάναμε και πολλά βήματα σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση πριν τι εκλογέ, Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε αργά το βράδυ κάποια συνεδρίασή μας πριν τις εκλογές, όπως θα θυμάστε. Έχουμε και τον υποπτικό μηχανισμό. Ε, θα αναλάβει δηλαδή σε δύο μήνες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα εποπτικές ε, αρμοδιότητες. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, βήμα, θα σπάσει ο σύνδεσμος μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη και όλα αυτά θα βελτιώσουν και το επενδυτικό κλίμα. Είναι πολύ σημαντικές <clears throat> οι συνεχιζόμενες ε, προετοιμασίες και όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι και εμείς θα εξετάσουν πολύ προσεκτικά τα επικαιροποιημένα, τις στοιχεία από την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και τις δοκιμές αντοχής, τα stress test. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, για την Τραπεζική Ένωση, τις συστάσεις ε, για την εξυγίανση των τραπεζών, έχουμε τις, ε, την οδηγία για την εξυγίανση και ανάκαμψη τραπεζών, έχουμε τον εννέο, μηχανι... μηχανισμό, τον μηχανισμό εξυγίανσης και όλα αυτά είναι προτεραιότητα και για την προτεραιότητα ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα τέλος να ολοκληρώσω αναφερόμενο στι χώρε οι οποίε εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομική προσαρμογή, Δύο είναι ε, προ το παρόν οι μόνο αυτέ που έχουν απομείνει, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Από την τελευταία φορά ε, που ήρθα στην Επιτροπή σα ε, βγήκε επιτυχώ από το μνημόνιο η Πορτογαλία χωρί όπω γνωρίζετε να ζητήσει περαιτέρω υποστήριξη. Η τελευταία τριμηνία αξιολόγηση του Κυπριακού Προγράμματο επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε τροχιά. Η Επιτροπή, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Τράπεζα συμφώνησαν τον Ιούλιο ότι η Κύπρος συνεχίζει να εκπληρώνει τους ε, δημοσιονομικούς της στόχους, υπάρχει σταθερή πρόοδος με την αδιάρθρωση των τραπεζών και συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις φυσικά απομένει μακρύς δρόμος, οπότε ε, το μόνο μπορώ να κάνω να τονίσω πόσο σημασία έχει η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση των ε, απαιτήσεων του προγράμματος. Το ε, Eurogroup θα εξετάσει τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης ε, της 12 Σεπτεμβρίου, στις 12 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα έχει γίνει πραγματική πρόοδος για την επαναξισορρόπηση της οικονομίας χάρη στις αξιοσημείωτες προσπάθειες που καταβάλουν και κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές αρχές επιδεικνύει πλέον πρωτογενές πλεόνασμα η Ελλάδα και η οικονομία της Ελλάδας ε, μετά από έξι χρόνια ύφεση ε, αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη το 2014. Έχουμε θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ε, ανακεφαλαιοποίηση του τομέα των τραπεζών και βλέπουμε να αυξάνει και η εμπιστοσύνη των αγορών. Παραμένουν όμως πολλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων το πάρα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος. Και επίσης, παρά το ότι φαίνεται να αρχίσει να μειώνει το 2014, παρά αυτή η ανεργία παραμένει πολύ σε πολύ σημαντικότερα ποσοστά, υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και ιδίως μεταξύ των νέων. Και αυτό πρέπει να είναι η μεγαλύτερη μα προτεραιότητα. Η τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο. Η, τέ, η πέμπτη αξιολόγηση θα λάβει χώρα το φθινόπωρο. Και στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης θα εξετάσουμε ποια μελλοντικά μέτρα ενδέχεται να χρειαστεί να υλοποιηθούν, καθώς θα, ε, επίσης θα αξιολογήσουμε και τις ε, μελλοντικέ ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας. Οποιαδήποτε απόφαση για το κατά πόσο θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση Ελλάδα μετά το τέλος του μνημονίου θα ληφθεί μετά την ε, αξιολόγηση και υπό το πρίσμα της αξιολόγησης. Αυτά έχω να πω μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για τι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις σας. Να ξεκινήσουμε τώρα το γύρο των ερωταπαντήσεων. Πρώτα απ' όλα ο συντηνιστής του ΕΛΚ, ο κ. Μπάλτς, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Ντέσιλμπλουμ. Χαιρόμαστε που ως πρόεδρος της Ευρωζώνης βρίσκεστε και πάλι εδώ μαζί μας στην Επιτροπή. Θα ήθελα να θίξω δύο θέματα, δύο περιπτώσεις. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη ομιλία του Μάριο Ντράγκη στο Jackson Hall, την οποία πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε, αλλά θεωρώ ότι επιδέχεται παρερμηνιών. Και αυτό έγινε στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτές τις παρερμηνίες αυτές, ο Μάριο Ντράγκη δεν έκανε ε, σύσταση για τέτοια πολιτική χρηματοδότησης και είναι σαφές ότι η καταπολέμηση της ε, ανεργίας προϋποθέτει αναγκαστικά μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές. Και η εκτίμηση των δημοσιονομικών, ε, γιατί είναι πολλέ οι κρατικέ δαπάνε ήδη σήμερα σε πολλά κράτη-μέλη και το μεγάλο φορολογικό φορτίο και οι, νομοθετικές, ε, οι νομοθετικοί περιορισμοί είναι αντίθετοι με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από δική σας πλευράς μια εκτίμηση για την ομιλία του κυρίου Ντράγκη γιατί θεωρώ ότι ανακοίνησε πολλά α, ε, αμφιλεγόμενα ζητήματα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο θέμα που ήθελα να θέξω. Το δεύτερο. Στην παρούσα φάση ε, καθημερινά αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίζουμε θέματα που αφορούν τη Ρωσία. Μας απασχολεί το θέμα αυτό καθημερινά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στη Ρωσία είναι τεράστια τα ποσά κεφαλαίου που διαφεύγουν. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς εκτιμάτε την κατάσταση στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ρωσία και κυρίως ως πρόεδρος της Ευρωζώνης. Πώς αξιολογείτε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις προοπτικές σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, τις περαιτέρω κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ρωσίας. Ευχαριστώ. The answer for the president is σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάλτση για τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες είναι και οι δύο αφορούν φλέγοντα θέματα. Όποια εφημερίδα και να ανοίξετε θα βρείτε σχόλια για τον Jackson Hall και για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Καταρχάς, το πρώτο θέμα, έχετε δίκιο. Οι ερμηνείες της ομιλίας ήταν ε, πολλές και διαφορετικές και πραγματικά ο καθένας επέλεξε ότι τον βόλευε ίσως. Άρα πάντα ε, είναι σόφρον να κοιτάξουμε την ίδια την ομιλία και να δούμε επακριβώς τι είπε ο κύριος Ντράγκη. Όντω λοιπόν ε, τόνισε ότι η χρηματοπιστωτική πολιτική θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό θεωρώ ότι συνάδει με, τα, με τις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα αυτό και γιατί πάντα ξεκαθάρισε ότι πολιτική δεν... Ε, ε ότι οι πολιτικοί δεν περιμένουν όλες τις απαντήσεις από τις τράπεζες και ότι οι τράπεζες δεν περιμένουν όλες τις απαντήσεις από τον χρηματικό κλάδο. Σε αυτό λοιπόν ήταν συνεπής και ξεκαθάρισε ότι το Σύμφωνο Ανάπτυξης και σταθερότητα αποτελεί μια άγκυρα εμπιστοσύνης. Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Και δεν θα μπορούσαμε να το καταρρύψουμε το σύμφωνο. Ο Μάριο Ντράγκη σε κάθε ομιλία υπογραμμίζει την σημασία των διορθωτικών αλλαγών σε ό,τι αφορά την βελτίωση εκβάθρων τη ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησατε για τη αγορά εργασία. Αυτό αποτελεί θέμα σε πολλές χώρες γιατί υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν πραγματικά διαφορετικές ανάγκες μεταρρυθμίσεων στι διάφορε χώρες. Σε ό,τι αφορά την χρηματοπιστωτική πλευρά, υπάρχουν διάφορες ε, εναλλακτικέ σε ό,τι αφορά το σύμφωνο και θεωρώ ότι είναι έντονη η δεσμεύση τη Ευρωζώνη στου κανόνε του σύμφωνου με την απαραίτητη ευελιξία όπου αυτή ενδείκνεται. Αλλά στη χρηματοπιστωτική πολιτική υπάρχουν διάφορε επιλογέ που μπορεί να κάνει κανεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία που συμπεριλαμβάνεται και προβλέπεται από τους κανόνες του συμφώνου και ύστερα υπάρχουν επιλογές πιο φιλικές προς την ανάπτυξη Εντό τη χρηματοπιστωτική πολιτική, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, μπορεί κανεί να προβλέψει ένα περιθώριο για την φορολογικό βάρο, για του φόρου επί τη εργασία, μετατοπίζοντα την φορολογική πίεση σε άλλου τομεί που έχουν ε, υποστεί λιγότερε ζημιέ ε, ή κάνοντα περικοπέ με πιο φιλικό προ την ανάπτυξη τρόπο. Ω εκ τούτου, δεν νομίζω ότι η συζήτηση για τη χρηματοδοτική πολιτική ε, θα πρέπει να περιοριστεί στο κατά πόσο θα πρέπει να βάλουμε φωτιά στο σύμφωνο. Το σύμφωνο θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία για την αξιοπιστία μας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μέσα στο σύμφωνο προβλέπεται ευελιξία και στη χρηματοδοτική πολιτική μπορεί κανείς να κάνει έξυπνες επιλογές σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Για το δεύτερο θέμα, για τη Ρωσία. Αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί ιδιαίτερα θέμα για την Ευρωζώνη. Θα μπορούσα λοιπόν να σταματήσω στο σημείο αυτό, να πω δύο λόγια παραπάνω ωστόσο. Θεωρώ ότι οι κυρώσει, ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, έχουν αποτέλεσμα. Αγγίζουν τον πυρήνα τη οικονομία στην Ρωσία ασφαλώ. Και θεωρώ ότι υπάρχει η επιλογή και θα ήταν ε, πραγματικά ενδεχομένως σωστή επιλογή να αυξηθούν οι κυρώσεις σταδιακά, βαθμιαία, όχι να κλιμακωθούν ε, υπέρμετρα. Θα πρέπει λοιπόν να ταχθεί η Ευρώπη υπέρ της υποστήριξης της Ευρώπης, της Ουκρανίας, συγγνώμη. Και οι οικονομικές κοινώσεις είναι σημαντικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, και τώρα να δώσω το λόγο στον Ούντο Μπούλμα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Ντέισελμπλουμ. Σας καλωσορίζω και από πλευράς των συναδέλφων από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών εδώ στην Επιτροπή μας. Ας μην ας αφήσουμε τις χειριτούρες. Η κατάσταση δεν είναι καθησυχαστική. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα τέλμα. Δεν είμαστε με το ένα πόδι στον κρεμό πλέον. Αλλά διακινδυνεύουμε να μείνουμε σε αυτό το τέλμα μακροπρόθεσμα. Κάπως θα πρέπει να βγούμε από το βούρκο το πόσο σημαντικό είναι το ότι παρενέβη και θα πρέπει να παρέμβει ο Μαρεντράγκη φαίνεται από το γεγονός ότι ο αξιότιμος συνάδελφος κύριος Μπάλτσε ξεκίνησε την εισήγησή του λέγοντας ότι αυτό που δεν θα μπορούσε να εννοεί σίγουρα ο κύριος Τράγκη με την ομιλία του, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύσαμε τα λόγια του. Α συζητήσουμε λοιπόν το πώς θα βγούμε, πώς θα εξέλθουμε, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να ερμηνεύσουμε την ομιλία του, το θέμα είναι τι θα κάνουμε, το θέμα δεν είναι... Δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν οι απαραίτητε αποταμιεύσεις και θα αποφέρουν κέρδη στα κράτη. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε πρόγραμμα για αυτό που είπε ο Ντράγκη. Ούτε πολιτική συνένεση, ούτε το πρόγραμμα για να εφαρμοστούν όλα αυτά που είπε ο Ντράγκη. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας κάνω μια επερώτηση σε ό,τι αφορά η ευελιξία. Από πού θα έρθει αυτή η ευελιξία. Φυσικά συζητάμε δικαίω για διαστατικές ε, μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την ροή των επενδύσεων, αλλά δεν είναι δυνατόν ο καλύτερος... Ε, η ο Υπουργό που επιτρέπει τι επενδύσει. Δεν μπορεί να παραγορεύονται οι επενδύσει στην Ευρώπη. Δεν απαγορεύονται οι επενδύσει στην Ευρώπη. Πού θεωρείτε ότι είναι η πολιτική βούληση, πού είναι τα προγράμματα. Δώστε μα κάποιε σύμβουλε για να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και με του υπουργού. Και πείτε μα ποιο είναι ο ρόλο του δημοσίου σκέλου. Πού μπορεί να δράσει ο δημόσιος τομέας για να καλέσει, να προσκαλέσει, να παροτρύνει και τους ιδιωτικούς ε, φορείς να κάνουν επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς που χρειαζόμαστε. Αυτό ερωτώ. σα ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω η προσέγγιση του να δούμε σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόμαστε τώρα θα πρέπει να βασιστεί σε μια ανάμειξη πολιτικών δεν νομίζω ότι εσείς οι πολιτικοί θα πρέπει τη μεριά σας να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας εργαλεία ή να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που λέει ότι όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να έρθουν από την Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει μια, σειρά, υπάρχει μια σειρά από αποκρίσει, κάποια συγκεκριμένα βήματα που έκανε η Κεντρική Τράπεζα ήδη από τον Ιούνιο. Θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτά και υλοποιούνται καθώ μιλάμε. Τα αποτελέσματα βέβαια δεν τα έχουμε δει ακόμη λόγου χάρη για το πρόγραμμα της Κεντρικής Τράπεζας για το LTRO θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα προχωρήσει του χρόνου και τους ερχόμενους μήνες περιμένουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Αλλά ήδη τον Ιούνιο κάποια πρόσθετα μέτρα ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα το πώ ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα δεν θα φανεί σε μία ή δύο εβδομάδε. Χρειάζεται χρόνο. Καταλαβαίνω την ανυπομονησία σα. Επίση, για την Τραπεζική Ένωση θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι αν τα πάμε καλά, εάν μπορέσουμε όντω να δώσουμε νέα μορφή στον τραπεζικό μα τομέα, θα πρέπει να δούμε πώς θα συμβάλλει και στην οικονομική μας ανάκαμψη η Τραπεζική Ένωση. Πιστεύω ότι είναι ένα καθοριστικό κομμάτι της στρατηγικής μας για να ξεκινήσει η ανάπτυξη πάλι στην Ευρώπη, να ξεκινήσουν οι επενδύσεις και ούτω καθεξής. Βεβαίως, προφανώς, οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη προτεραιότητα στον κατάλογο πατριωτήτων μας, περισσότερο από ό,τι πριν από ένα εξάμεινο, αλλά ακόμη προσπαθούμε και περιμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο από τις αποφάσεις για το πακέτο εποπτείας του Ιουνίου, και εν καιρό θα ξέρουμε ακριβώ τι θα γίνει με τις επενδύσεις. Τα 300 δις ε, που αναφέρθηκαν ε, ως στόχος ήταν ε, πραγματικά μία αναφορά που έγινε θερμά δεκτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη της τις προτεραιότητες αυτές, τους στόχους αυτούς για να προχωρήσει και για την ευελιξία θα πρέπει στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο να την χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε, χωρίς όμως την αξιοπιστία στην οποία έχουμε συμφωνήσει να την διαταράξουμε. Η ευελιξία δεν σημαίνει ότι, μπορεί να γίνει, ότι τα πάντα μπορεί να ισχύουν. Ευελιξία θα πει ότι πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές προσπάθειες, διαρθρωτικές βελτιώσεις. Επίσης μπορεί να σημαίνει ευελιξία ότι θα λάβουμε υπόψη τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις διάφορες χώρες. Βάσει μια τέτοιας αποτίμησης και εφόσον αντιμετωπιστεί το διευθυντικό έλλειμμα, εφόσον υπάρξουν βελτιώσεις εκεί, ε, εφόσον μια σειρά από διευθυντικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν, τότε η ευελιξία θα μπορεί να ε, χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συζήτηση αυτή όμω θα γίνει πιο συγκεκριμένη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν θα έχουμε τα πρώτα σχέδια προπολογισμών ε, και την αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευελιξία λοιπόν μεν, αλλά όχι ε, ό,τι λύση να είναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο. Και τώρα για τους θετικούς και ο κ. Μαριάς δεν θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις που κάνατε τόσο για τη γενική οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια και τα εκατομμύρια των ανέργων και η φτωχοποίηση στην Ευρώπη δείχνει ότι έχει αποτύχει η πολιτική και η πολιτική που κάνετε στο Eurogroup αλλά και για την Ελλάδα. Να σας επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέχρι σήμερα 214 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια επί τέσσερα χρόνια και όμως έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, η ανεργία των νέων έχει φτάσει στο 53%, χιλιάδες μαγαζιά έχουν κλείσει, το 40% του ελληνικού λαού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, το ΑΕΠ έχει μειωθεί 25%, το δημόσιο χρέος έχει ξεφύγει και είναι πλέον μη διαχειρίσιμο αφού από 125% έχει φτάσει στο 178% τα κόκκινα δάνεια που οφείλουν οι ιδιώτες σε τράπεζα στα 60 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν η πολιτική σας στην Ελλάδα έχει αποτύχει. Και αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που λέτε ότι υπάρχει, πρώτα απ' όλα υπάρχει για να πληρωθεί σύμφωνα με το μνημόνιο το κεφάλαιο των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα και δεύτερον προέκυψε από τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ, σας τα λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο με απόφασή του το Μάρτιο απέδειξε ότι έχετε τεράστιες ευθύνες και εσείς ως Eurogroup που κατευθύνετε την πολιτική της Τρόικας και η ίδια η Τρόικα. Και αναγράφονται συγκεκριμένα οι ευθύνες για την έλλειψη πρόβλεψης των κοινωνικών επιπτώσεων του προγράμματος προσαρμογής, για το λάθος πολλαπλασιαστή, για τη μείωση των συντάξεων. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και απλά ως προς την ερώτηση που θα κάνω. Πρώτον, προτίθεστε ως eurogroup να αποζημιώσετε την ελλάδα για την τεράστια οικονομική ζημιά την οποία έχει υποστεί. δεύτερον ποιο είναι το follow up αυτής εδώ της απόφασης του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την οποία την άλλη εβδομάδα θα στείλω επιστολή στους συναδέλφους για να προχωρήσουμε διότι σε αυτή την απόφαση γράφεται ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα του χρέους. Πρέπει να κουρευτούν κατά την άποψή μας τα ομόλογα της Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να διαγραφεί μεγάλο μέρος του χρέους. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αλλά και το σημείο του 72 της έκθεσης αναφέρει ότι πρέπει να γίνει διευθέτηση του χρέους. Πιστεύετε σωστά ότι η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη το 2014 όπως μας είπατε. Ποια είναι τα στοιχεία, από πού προκύπτει. Ήδη δεν έχει ανάπτυξη τώρα. Θα συνεχίσετε στο Παρίσι που γίνονται τώρα οι διαπραγματεύσεις της Τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση να ζητάτε να υπάρξουν νέες απολύσει, να μην υπάρξει προστασία πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, να μην υπάρχουν φοροαπαλλαγές, να μην μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και κρυώνει όλος ο ελληνικός λαός κάθε χρόνο. Θα συνεχίσετε λοιπόν αυτή την πολιτική. Um, uh, Νομίζω σε περασμένε συνεδριάσει τη Επιτροπή σα και σε συναντήσει μα συχνά συζητήσαμε το θέμα τη Ελλάδα. Κανεί δεν διαφωνεί για το πώ έχει κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ήταν σοβαρότατο ο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο για όλο τον ελληνικό λαό και πολλά από αυτά που είπατε είναι αλήθεια. φτώχεια, ανεργία. Αλλά φαίνεται να το διασυνδέεται αυτό με το πρόγραμμα. Νομίζω ότι τα αίτια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δεν ήταν το μνημόνιο ή το πρόγραμμα της Τρόικας. Ήταν ε, μακροχρόνιο το πρόβλημα και οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Αυτή την ε, μελέτη όμως θα πρέπει να την κάνουμε σε μια άλλη φάση. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πολλά από τα διαρθρωτικά προβλήματα που ανέκαμψαν ή αναχέτησαν την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του μνημονίου. Δεν υπάρχει απλή λύση. Διότι αν θέλουμε να αλλάξει η βασική δομή μια οικονομία, να γίνει πιο ανταγωνιστική, να επιστρέψουν οι επενδυτέ στη χώρα, τότε χρειάζονται πραγματικά ευάθρων αλλαγέ. Δεν υπάρχουν ε, δυστυχώ ε, ε, τρόποι να αλλαξει η βασικη δομη μια οικονομια να γινει πιο ανταγωνιστικη να επιστρεψουν οι επενδυτε στη χωρα τοτε χρειαζονται πραγματικα βαθρων αλλαγε δεν υπαρχουν δυστυχω τροποι να πάρει κανείς την παρακαμπτήριο εδώ και να βρει λύσει. Όμως, ε, όπως και προηγουμένως, θα σταθούμε στο πλευρό της Ελλάδας ως Ευρωπαίοι εταίροι, θα τη στηρίξουμε όποτε χρειαστεί και αυτό βάσει της αναθεώρησης που τώρα θα ξεκινήσει. Μιλήσατε για το Παρίσι. Ξεκινάει η πέμπτη αναθεώρηση. Η πέμπτη μάλλον φάση αξιολόγηση και εκεί θα δούμε τι περαιτέρω βοήθεια μπορεί να χρειάζεται, τι περαιτέρω στήριξη μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου. Έτσι κι αλλιώ υπάρχει μια ατζέντα ανάπτυξη στη συνεργασία μα με την Ελλάδα και υπάρχει και από την ελληνική πλευρά ε, με τη συμμετοχή των ε, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεργαζόμαστε στενά με την ελληνική κυβέρνηση πάντως για όλους αυτούς τους σκοπούς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα για τους φιλελεύθερους, ο κύριος, η κυρία Φανχόιζεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντάισελμπλουμ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω σε μια διαφορετική θέση πλέον και μπορούμε να συζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ατζέντα. Θα ήθελα να θίξω δυόμιση ζητήματα για την ακρίβεια, διότι δεν ξέρουμε και κατά πόσο θα παραμείνετε στη θέση αυτή και για πόσο καιρό. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα έχει να κάνει με την ε, διευκόλυνση την ποσοτική χαλάρωση. Η χαλάρωση είναι μια ιδιαίτερη ε, έννοια ούτως ή άλλως. Υπάρχει ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού σε σχέση με το χαμηλό πληθωρισμό που έχουμε τώρα. Είναι χαμηλές και τιμές της ενέργειας, κάτι που δεν είναι απαραίτητα αρνητικό και οι χαμηλές τιμές των τροφίμων. Ως Eurogroup, ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος εδώ και τι ακριβώς θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά και ανάπαλη. Επίσης υπάρχει η έννοια της ελαστασφάλειας, δηλαδή μια ε, ισορροπία, ένα σημείο ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας σε σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τις ε, αναχώρα συστάσεις έγινε πολλή συζήτηση για το θέμα αυτό της ευελιξίας. Συμφωνείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ και το θέμα της ασφάλειας, διότι είναι πολλές οι χώρες που ακόμη δεν συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, ούτε ε, συμμορφώνονται πλήρως με τις αναχώρα συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι που σας, είδα, που σας βλέπω εδώ, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά. Είσαστε πρόεδρος της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και άρα συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στην Χάγη. Για την πρώτη σας ερώτηση, για το κατά πόσο θα μείνω στη θέση αυτή και για πόσο. Ε, χαίρομαι που θέλετε την ερώτηση αυτή. Όπως θα ξέρετε, αλλά ευχαρίστως να μοιραστώ αυτή πληροφορίες και με άλλους, η θητεία μου ε, λύγει τον Ιούλιο του επόμενου έτους. Και είμαι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη θητεία μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσω πιο νωρί. Και μετά θα, υπάρξει υποψήφι, θα υπάρξουν υποψήφοι και θα ληφθεί απόφαση για την επόμενη θητεία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε λιγότερο, να συζητάμε λιγότερο την ε, δουλειά των πολιτικών μας και πιο πολύ τη δουλειά των, του εκλογικού μας σώματος, των περιφερειών μας. Για, το, για την προσωπική χαλάρωση. Σας απασχολεί ο όρος χαλάρωση. Η προσωπική χαλάρωση, το QE, μπορεί να είναι ένα καλό εργαλείο ανάλογα με την ερμηνεία σας γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρευστότητα στην αγορά και το, το ερώτημα είναι κατά πόσον όλα τα μέσα τα οποία έχει εκδώσει η ΕΚΤ αρκούν για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από την κρίση της ΕΚΤ και εγώ πιστεύω πραγματικά είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να υπάρχει εξαρτησία της ΕΚΤ και όπως σας είπα το πακέτο του Ιουνίου δεν έχει εξεταστεί ε, αρκετά στις αναλύσεις μας και τα αποτελέσματα του πακέτου Ιουνίου και σε ό,τι αφορά το LTRO, τη μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνουν πιο επισταμένα. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι αυτό επαφείται στην ΕΚΤ. Το ίδιο ε, ισχύει και για τον κίνδυνο πληθωρισμού σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Μιλήσατε για την, ε, το flexicurity, αυτή την ευέλικτη ασφάλεια. Αυτό χρησιμοποιείται συχνά ως όρος και στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Και μιλήσατε για τα πακέτα, τι γίνεται με τον τομέα της ε, ευελιξίας, εντάξει, με τον τομέα της ασφάλειας, τι γίνεται, είπατε. Αυτό εξαρτάται από τη σημασία των συμφώνων. Αυτό δεν θα πρέπει να το υποτιμάμε και αυτό το είπε και αρκετά ρητά ο Μάριο Ντράγκη στην ομιλία του Τούτου λεχθέντο, ωστόσο, θεωρώ ότι η ευελιξία έχει μπει στην, στο όλο για κάποιον λόγο. Αποτελεί έναν όρο, μία προϋπόθεση. Και αυτή η ευελιξία μπορεί να υπάρχει μόνο υπό συγκεκριμένου όρου. Και αυτό λοιπόν διευκρινίζεται. Και έχει άλλωστε χρησιμοποιηθεί. Αν κοιτάξετε τι γίνεται και πω εφαρμόσαμε του χρηματοπιστωτικού κανονε και τη σχετική πολιτική τα τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι Διάφορες χώρες έχουν λάβει πιο πολύ χρόνο υπό συγκεκριμένους όρους. Ενίοτε, για παράδειγμα, οι 100 χώρες είχαν λάβει πιο πολύ χρόνο αρκεί να υπήρχε στη συνέχεια ονομαστικό πακέτο. Ήταν και αυτό λοιπόν μια δυνατότητα, μια άλλη δυνατότητα που είχα ζητήσει εγώ ήταν αν οι χώρες ζητούν πιο πολύ χρόνο και αυτό πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πακέτο από συγκεκριμένες διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Αν δηλαδή αξιώνουν πιο πολύ χρόνο και έχουν δικαίωμα σε πιο πολύ χρόνο για να πετύχουν τους του στόχους, θα πρέπει να φροντίσουμε ο χρόνος αυτός να αξιοποιείται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιείται ο χρόνος αυτός για να γίνονται ε, μεταρρυθμίσεις. Ο Φάμπιο Ντεμάζη από την ΚΟΕ τώρα λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Παρακαλώ να με συγχωρήσετε για την νομή, και το, μη, όχι τόσο κοινοβουλευτική μου γλώσσα, αλλά εάν ε, ανακεφαλαιώσω την, ε, ε, το συμπέρασμα της έκθεσής σας, αυτό που λέει είναι ότι είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, τα έχουμε πάει χάλια και πρέπει να να βρούμε μία λύση. Από την Ιταλική μου κουλτούρα, τι να σας πω, ξέρω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές θυσίες και ότι αυτό που αναμένουμε πλέον είναι μια λύση στον παράδεισο, τίποτε παραπάνω. Η όλη η ιστορία με την Τρόικα μας λέει ότι αν σφίξουμε το ζωνάρι και αν κάνουμε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ε, μπορεί να βγούμε από το τέλμα. Οι Ευρωπαίοι μας ρωτάνε πότε, πότε θα γίνει όλο αυτό. Ε, ήδη ε, βλέπουμε να έχουμε χάσει μια δεκαετία στην Ευρώπη και εγώ όταν ε, ήμουν στο σχολείο δίδασκα στους ε, μαθητές μου ότι μπορείτε να προβάλλετε ό,τι επιχείρημα θέλετε θεωρητικά και να είσαστε και υπέρ ή και κατά της λιτότητας, αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα και πραγματικά δεδομένα βασισμένα στην πραγματικότητα. Ε, τα πραγματικά αποτελέσματα μας λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιαπωνία, όποιος είναι εκτός ευρωζώνης τα πάει καλύτερα από εμά. Ε, το ΑΕΠ έχει αυξηθεί ε, σε άλλες χώρες, αλλά όχι στις χώρες ε, του Μονίου ή στην Ιταλία που έχει μειωθεί. Η Ισπανία λίγο τα πάει καλύτερα, αλλά η δημοσιονομική μόχλευση για όσους δεν κατέφυγαν στην λιτότητα και περιόρισαν απλώ τι δαπάνε του, ήταν μια καλύτερη λύση. Διαβάζοντα λοιπόν την εκθεσή σα, διαρωτώ με, η αναχώρα συστάσει γιατί δεν κάνουν καθόλου λόγο για την παραβίαση των μακροοικονομικών στόχων. Δεν κάνουν καθόλου λόγο για τους στόχους πληθωρισμού που ε, προσεγγίζει αλλά είναι κάτω από το 2% και εδώ δεν επιτυγχάνουμε σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά γι' αυτό στην έκθεσή σα. Νομίζω ότι είναι μια βασική παραβίαση καθοριστικών μακροοικονομικών στόχων τη Ευρωζώνης. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε, ε, επειδή είναι τόσο ε, ε, πεπισμένη η γερμανική κυβέρνηση, ότι πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ δεν είμαι δογματικό εδώ. Αλλά πώ βλέπετε το τηλεφώνημα τη κυρία Μέρκελ και του κυρίου Ντράγκη που τον πίεσε να συνεχιστούν οι πολιτικές λιτότητας. Και κατά δεύτερον, πώς βλέπετε την αναγγελία ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αγοράσει και πάλι ομόλογα. Με τον εκφρασμένο στόχο ότι αυτό θα δώσει πάλι ε, χρήμα για την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Η ερώτησή σα για το τηλεφώνημα που έλαβε ή δεν έλαβε χώρα είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν ήμουν παρόν, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αυτό που πιστεύω ωστόσο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποδείξει ότι είναι, ένας, ότι είναι μια πολύ ισχυρή κεντρική τράπεζα. Μεγάλη σημασία για την Ευρωζώνη καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Νομίζω ότι η προσέγγιση τους και τα εργαλεία που έχουν ως τώρα δείξει ότι διαθέτουν ήταν πολύτιμα και θα γίνουν ακόμα πολύτιμότερα το ερχόμενο δίμηνο. Υπάρχει βέβαια το θέμα του κατά πόσον τα εργαλεία αξιοποιήθηκαν πλήρως. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι έγινε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και όλες τις λύσεις από την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέτε όλοι τα πάνε καλύτερα εκτός Ευρώπης και εκτός Ευρωζώνης. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι η ίδια μας η νομισματική πολιτική ενέχει πολλούς κινδύνους που μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην υλοποιηθούν, να μην λάβουν σαρκοκιωστά, αλλά θα μπορούσαν στο μέλλον να, και θα έπρεπε στο μέλλον να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που μπορεί να προέρχονται από την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ λόγω χάρη. Και ο αντίκτυπο γίνεται αισθητό σε, διεθνέ επίπεδο και στι νέε οικονομίε. Μην περιμένουμε λοιπόν όλε τι λύσει από την νομισματική πολιτική. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη, τη θητεία και το, την αρμοδιότητά τη για να κάνει όσα είναι αναγκαία. Στην Ευρώπη όμω, κατά τα άλλα, πιστεύω ότι κάποιε χώρε έχουν περισσότερο δημοσιονομικό περιθώριο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ε, το επίπεδο των ε, δημόσιων επενδύσεων σε κάποιε χώρε θα μπορούσε να αυξηθεί. Λόγω χάρη για τι υποδομέ. Νομίζω ότι σε ορισμένου τομεί τη οικονομία, σε ορισμένε χώρε υπάρχει περιθώριο για την μισθολογική βελτίωση. Αυτό θα μπορούσε να τονώσει να επιταχύνει την ανάκαμψη της ε, ζήτησης. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, συγκεκριμένοι στο τι ισχύει και συμβαίνει σε κάθε χώρα, στην ανταγωνιστικότητα ορισμένων τομέων της κάθε χώρας. Πρέπει να είμαστε πραγματικά ε, πολύ συγκεκριμένοι στις λεπτομέρειες για να βρούμε την κατάλληλη, το κατάλληλο μείγμα πολιτικών που χρειάζεται. Αλλά σίγουρα εδώ θα παίξουν μεγάλο ρόλο οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις και η βελτίωση ε, των μισθών σε πολλούς τομείς τη οικονομία. Θα πρέπει να υπάρξει ανάμειξη πολιτικών λύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μέχρι τώρα φανήκαμε ελαστικοί στην ε, χρήση του χρόνου, αλλά τώρα θα πρέπει να παραμένουμε πολύ πιστοί στου κανόνε. Ιδάλω δεν θα έχουν χρόνο όλοι οι συνάδελφοι για να μιλήσουν. Γι' αυτό παρακαλώ θέμα του συναδέλφου να μην θέτουν ερωτήματα τριών και τρισήμιση λεπτών για να μπορέσουν και ο προσκεκλημένος με τις απαντήσεις του να παραμένει στα πλαίσια του πενταλέπτου. Ιδάλλως κάποιοι συνάδελφοι δεν θα λάβουν το λόγο. Επόμενος, για τους πράσινους, ο κ. Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεσεμπλόμου. Είπατε ότι είμαστε πιο αυστηροί, ενδιαφέρον. Για... Ε, κύριε Πρόεδρε, όμως να είστε λίγο πιο δικαιοί. Ε, κύριε Ντέσσερμπλουμ, καλώς ορίσατε. Ούντο, δεν ξέρω τι αίσθηση έχεις εσύ, αλλά ε, με ένα σοσιαλιστή σαν τον Ντέσσερμπλουμ, ποιος χρειάζεται τους θρεπτικούς, γιατί κύριε Ντέσσερμπλουμ, λυπάμαι, αλλά αυτά που είπατε θα μπορούσατε να τα έχει πει ο κύριος Ντεγκίνδος ή οποιοδήποτε άλλος. Εγώ Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τα φαινόμενα και τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Αποτελέσματα τα οποία θα έπρεπε να σας μιλήσουν στην καρδιά. 25% του κόσμου με, σε φτώχεια, σε κοινωνικό αποκλεισμό σχεδόν. Έχετε δίκιο λοιπόν, έχουν αποτελέσματα οι μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη που είναι ο στόχος σας. Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Αν είναι λοιπόν κανείς υπεύθυνο ηθήνων, θα πρέπει να έχει και ένα σχέδιο Β. Ποιο είναι το σχέδιο Β λοιπόν, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ποιο είναι το σχέδιο Β, εάν ε, δεν μειωθεί η ανισότητα, το οικολογικό αποτύπωμα που μάλλον δεν σας απασχολεί. Μιλήσατε για φορολογική μετατόπιση, όλοι συμφωνούν. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά τι άλλο θα έπρεπε να ε, φορολογηθεί, γιατί πρόκειται για μετατόπιση. Αν δεν φορολογηθεί ο ένας, ποιος θα φορολογηθεί. Και τέλος, πείτε μου με ναι ή όχι, το κοινοβούλιο αυτό έχει εργαστεί ε, σε ό,τι αφορά ανάλυση του έργου της Τρόικα. Είμαι βέβαιος ότι θα υποστηρίξετε μια επίσημη έρευνα του έργου της Τρόικα προκειμένου να είναι καλύτερα το μελλοντικό της έργο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε ότι οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε φτώχεια. Αυτό είναι ενδιαφέρον ως ε, παρατηρήση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι την κατανοώ απόλυτα. στη δική μου τη χώρα και μιλώ τώρα ως Ολλανδός ε, υπουργό, κάναμε και κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, επανήλθε η ανάπτυξη κοιτώντας χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιρλανδία, ελήφθησαν σκληρά μέτρα. Έγιναν μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές αγορές και πραγματικά επανήλθε ένας ρυθμός ανάπτυξης. Μου φαίνεται ότι στην ανάλυση της κρίσης αυτής έχουμε την τάση να κατηγορούμε τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν πρόσφατα για κάποια από τα εγγενώς διαρθωτικά ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στην ε, οικονομία μας και αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά η ανεργία των νέων για παράδειγμα θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί αν θέλουμε να έχουν ευκαιρίες οι νέοι στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ανοίξουμε την αγορά εργασίας. Αν θέλουμε να έχουν καλύτερες ευκαιρίες για να βρουν μια δουλειά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι, ότι θα έχουν δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τα επαγγέλματα αυτά. Αυτό λοιπόν προαπαιτεί μεταρρυθμίσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λύση να αποδεχτούμε στις οικονομίες μας το χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και μετά να περιμένουμε ότι θα επανέλθει η ανάπτυξη. Ούτε πιστεύω ότι όλες οι απαντήσεις θα έρθουν από το δημόσιο τομέα και από τις δημόσιες δαπάνες. Δεν είπα ότι το είπατε εσείς αυτό, απλά σας λέω ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει καλό μείγμα πολιτικών και θα πρέπει να προσαρμόζεται στον δρόμο αυτή η πολιτική και θα πρέπει να κοιτάξουμε την ατζέντα επενδύσεων. Πώς θα προσελκύσουμε υψηλό επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία στο χρηματοπιστωτικό σύμφωνο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες της νομισματικής πολιτικής με σωστό τρόπο εντός της εντολής της τράπεζας και έτσι θα σχηματίσουμε αυτό το μείγμα των πολιτικών των πολιτικών. Αλλά μην το κάνετε. Και εγώ δεν πρέπει να το κάνω. Ότι αν μείνει η κατάστασή όσο έχει και θα δαπανίσουμε πιο πολύ χρήματα, θα επενδύσουμε και θα βγούμε από την κρίση. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία. 30 δευτερόλεπτα έχω ακόμα, λέει ο κ. Λαμέτ. Δεν το είπα αυτό, απλά σημειώνω ότι είπατε ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας που είναι πολύ χαμηλό, αλλά δεν είπατε τίποτα για την επίπεδο ανισότητα και φτώχεια, αλλά πολύ απλά δεν υπάρχει πρότυπα. Αν θέλετε να δείτε τι γίνεται, πήγετε στην Ιρλανδία, πήγετε στην Ελλάδα. Και αν δεν έχετε πάει ποτέ, βγείτε και δείτε τι γίνεται στους δρόμους. Ναι, το έκανα, απαντάει ο κύριος Ντέισελμπλουμ και θα το ξανακάνω. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι το να αντιμετωπίσουμε θέματα ανταγωνιστικότητας δεν είναι κάτι εγγενώς αντίθετο με την αντιμετώπιση των ανισοτητών και της, του κοινωνικού αποκλεισμού. Θεωρώ ότι το θέμα της ανταγωνιστικότητας αποτελεί το, τη βάση για την ανάκαμψη, για την ανάπτυξη και μην δημιουργείτε τεχνητέ αντιφάσει. Ευχαριστώ για το FTT, ο Στίβεν Μούλερ. Good morning, Mr. Thank you. Καλημέρα σα, σα ευχαριστώ κύριε Ντέζελ. Σα ευχαριστώ για την ενημερωτική αναφορά που μα κάνατε. Μα ενθαρρύνει το γεγονό ότι εδώ μιλάμε για τη φτώχεια, τον πόνο, την οδύνη του λαού. Είπατε επίση ότι υπάρχει απώλεια ορμή ρυθμού, ιδίω των μεγάλων οικονομιών τη Ευρώπη, όπω η Γερμανία που φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ε, στο εμπορικό ε, σκέλος. Βλέπουμε τώρα ε, για τις κυρώσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να εφαρμοστούν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ε, άλλες ε, δικαιολογίες για το πού οφείλεται η κρίση, η κακή αγγλοσαξονική θεσμή, οι χώρες που δεν μπορούν να διαχειριστούν τις οικονομίες τους, η Ουκρανία τώρα με τις κυρώσεις κτλ. Όμως ε, δεν είναι αυτή η λόγια, αλλά είναι η πολιτική των θεσμικών οργάνων, η προηγούμενη και η τωρινή και δημιουργεί ε, θεσμικά προβλήματα. Πώς θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε αυτά. Επίσης, ο κύριος ε, Πάντοβαν, ο Ιταλός Υπουργό Οικονομικών, σε ένα πρόσφατο διάλογο συζήτησε το γεγονός και είπε ότι τρία χρόνια θα χρειαστεί μέχρι ότου βελτιωθεί η οικονομία μετά από τις μεταρρυθμίσεις. Στις μεταρρυθμίσεις σας λοιπόν, τις αλλαγές που προτείνετε, ε, τι θα γίνει, θα βοηθηθεί η κατάσταση των ανθρώπων, θα βελτιωθεί η ζωή του σήμερα. Υπάρχει επίσης έντονος αποπληθωρισμός, 0,6%. Και δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο την κατάσταση αυτό. Ούτε στη δική σας ανάλυση, ούτε σε άλλους αιματοπιστωτικούς οργανισμούς βλέπουμε κάποια στοιχεία βελτίωσης. Μόνο για το μακροπρόθεσμο ε, μέλλον μιλάμε, αλλά αυτό δεν βελτιώνει σήμερα τη ζωή του κόσμου. Επίσης, χαίρομαι που λέτε για, μιλάτε για το υψηλό μη μισθολογικό κόστος εργασίας και φυσικά και συμφωνούμε, αλλά τα σχόλιά σας για τις βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να, ε, εφαρμοστούν, αυτό είναι ανησυχητικό για μένα. Ψηφίστε να στηρίξετε τη φορολόγηση ε, των δημοσιονομικών ιδρυμάτων από την πίσω πόρτα. Μήπως προνείστε τα σχόλιά σας στην άποψη ότι θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο ε, της φορολόγησης των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα μας πείτε, θα δηλώσετε ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ποτέ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Δύο-τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα για την Ουκρανία. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πρώτα απ' όλο ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δεν προέκυψε ούτε χθε ούτε προχθέ. Αλλά από τότε που ε, υπήρξε κρίση στην Κρυμαία. Και τότε μπήκε στην ημερήσια διάταξη και τη δική μα και έκτοτε η κατάσταση επιδεινώνεται. Έχουμε πρόβλημα με τι επενδύσει, ε, με την κατανάλωση και αυτό πραγματικά επηρεάζει την οικονομία μας επηρεάζει επίσης πραγματικά και όσες επιχειρήσεις έχουν ε, εμπορική δραστηριότητα με την Ουκρανία και βέβαια και με τη Ρωσία και θα πρέπει να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Επίσης μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις που θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσουν και αυτό είναι αλήθεια. Μεταρρυθμίσεις και στο φορολογικό μείγμα, στη φορολογική πολιτική μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, ορισμένες εξ αυτών. Κάποιες άλλες χρειάζονται περισσότερο χρόνο, παραδείγματος χάρη αγορά κατοικίας Πολλέ φορέ η αγορά κινήτων χρειάζεται χρόνια για να ορθοποδήσει. Το ίδιο ισχύει για τις, αγορά, για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη όταν μελετούμε του στόχου για τα ελλείμματα, τα διευθυντικά ελλείμματα. Ξέρουμε ότι χρειάζεται χρόνο για τη βελτίωση των προπολογισμών. Και σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη το ότι οι μεταρρυθμίσει είναι μακροπρόθεσμε. χρειάζεται χρόνο για να αποδώσουν. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Και όταν θα αξιολογήσουμε το 2-pack και το 6-pack, ε, θα τα λάβουν υπόψη και έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτά τα δύο πακέτα μέτρων. Επίσης είπατε ποια είναι η δική μας ε, δουλειά για το φορολογικό, για τη φορολογική πολιτική στην Ευρωζώνη. Μην ανησυχείτε. Πρέπει να αναλύσετε τις φορολογικές, τα φορολογικά ισχυρά και δύνατα σημεία των χωρών. Είπα ότι έχουν πολύ ψηλό μείνει στο λογικό κόστος σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό είπα. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Γίνονται πολλά στι ε, κάτω χώρες, στην ε, Ισπανία, στη Γαλλία. Υπάρχουν πολιτικέ πρωτοβουλίε για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε πόσο επίγον είναι, πώ πρέπει να γίνει, να μην γίνει αν ε, μετακυλήσουμε την ε, φορολογική πίεση σε άλλου τομεί, πώ θα γίνει αυτό ώστε να ε, είναι όσο το λιγότερο επιζήμιο αυτό για την οικονομία και ούτω καθεξή. Σημαίνει αυτό τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει τα ενία τη φορολογική πολιτική. Όχι. Μιλάμε εδώ για συντονισμό των πολιτικών. Όμω, θεωρώ και κατά ψευδόντα δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να συζητούμε περισσότερο για το συντονισμό των φορολογικών πολιτικών. Φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, και ούτω και διάβρωση της βάσης ε, και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και είναι και ένα κομμάτι της στρατηγικής μας για να ενισχύσουμε τη βάση της οικονομίας μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Μπερνάρ Μονό για τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω εκπρόσωπο των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωζώνης ένα ερώτημα έχω να σα υποβάλω, αλλά με ανησυχεί η ανικανότητα στην Ευρώπη για ανάκαμψη, για νέε θέσει εργασία, αλλά και γιατί δεν θέτει η ηγεσία της Ευρώπης ε, τα σωστά ερωτήματα. Στο δημοψήφισμα του Μάστρια το 1992 οι Γάλλοι ε, πολιτικοί θύνοντε και σε άλλε χώρε είχαν υποσχεθεί πλήρη απασχόληση, ευημερία. 20 χρόνια μετά πού βρισκόμαστε όλοι κοινωνικο οικονομική δείκτες είναι στο κόκκινο, έχουμε ενδυμική ανεργία σε όλες τις ε, τάξεις, τις ηλικιακέ, έχουμε κίνδυνο διαφρωτικής ύφεση και αποπληθωρισμό όπως ακούμε σε όλα τα πολιτικά σχόλια και στον τύπο. Μείωση τη ανταγωνιστικότητας, ε, και η Γαλλία έχει μπει στο στάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο εκτός της ε, Γερμανίας, φορολογικά έσοδα πολύ λίγα, άρα χρειάζεται δρακόντια, ε, δρακόντια λιτότητα για όλους. Όμως πράσινοι όλοι οι δείκτες, οι θετικοί δείκτες οι δημοσιονομικοί μετά τη διάσταση του 2008 Βέβαια έχουμε μόνιμη ε, διάσωση και στήριξη των τραπεζών. Το χρηματιστήριο ανεβαίνει. Αλλά όλα αυτά πραγματικά είναι ανήθικα σε σχέση με την οδύνη και τις θυσίες των πολιτών. Είναι ανησυχητική κατάσταση, αλλά είναι αντικειμενική. Εσείς πιστεύετε ότι το άκρος φιλελεύθερο αυτό μοντέλο της Τρόικας για όλο και περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και για την ενοποίηση τραπεζών, ε, ίσως αύριο και, και νομισμάτων και ίσως και των συνταξιδοτικών συστημάτων. Είναι το καλύτερο μικροοικονομικό μοντέλο αυτό προς το γενικό συμφέρον των πολιτών. Εγώ είμαι υπέρ του μοντέλου του οικονομικού πατριωτισμού και φοβούμε ότι ο λαός που είναι αγανακτισμένος θέλει να αλλάξετε άρδιν πολιτική. Απλά ελπίζω αυτό να γίνει με δημοκρατικό τρόπο. Ευχαριστώ. Σε πολλά από αυτά που είπατε δεν θα συμφωνούσα. Αλλά το δίλεπτο που μου έμεινε θα αποφύγω να απαντήσω και κατά λεπτό ούτως ή άλλως. Θα επικεντρωθώ απλώ στην ιδιωτικοποίηση όπου σταθήκατε και αν ακολουθούμε την ορθή πορεία με τις ιδιωτικοποίησεις. Σε καμία περίπτωση χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα μνημονίου ε, δεν είναι το βασικό σκέλος οι ιδιωτικοποίηση. Οι προσδοκίες μας όπως αυτό το σκέλος των προγραμματών δεν είναι πολύ ψηλές και δεν είχαμε και εντυπωσιακά αποτελέσματα ως τώρα έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, συμπεριλήφθησαν στα διάφορα προγράμματα διότι υπήρχαν τέτοια επίπεδα χρέους σε κάποιες χώρες που έπρεπε να προβλεφθεί ε, ως ένα μέρος της λύσης και η ιδιωτικοποίηση κάποιων τομέων. Όμως τα αποτελέσματα ως τώρα δεν ήταν ε, και καταπληκτικά. Τώρα, εάν η συνολική προσέγγιση της Τρόικας είναι σωστή, Εάν σκεφτείτε ότι η προσέγγιση της Τρόικας είναι, ταυτίζεται με το Eurogroup, θα πρέπει να καταλάβετε ότι η Τρόικα δεν αποφασίζει μόνο τη, δεν σχεδιάζει τα προγράμματα λιτότητα. Ε, τα προγράμματα αυτά είναι αντικείμενα διαπραγμάτευση με τι ε, ενδιαφερομένε χώρε και μετά στο Eurogroup λαμβάνονται οι αποφάσει από του υπουργού όλων των χωρών. Οπότε αυτή η ιδέα ότι η Τρόικα από μόνη τη είναι σαν ανεξάρτητο φορέα, ανεξέλεγκτο, χωρί καμία δημοκρατική λογοδοσία και λαμβάνει αποφάσει, δεν ισχύει. Εάν θέλετε να επικρίνετε την Τρόικα, να επικρίνετε το Eurogroup. Διότι εμεί λαμβάνουμε τι αποφάσει, τι τελικέ για τα προγράμματα λιτότητα. Τώρα, εάν είναι σωστά, ε, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κάποια αποτελέσματα έχουν φέρει, διότι κατάφεραν να απομακρύνουν τι χώρε από το χείλο τη χρεοκοπία, αλλά Εάν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ή θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τα πράγματα διαφορετικά, ίσω. Ίσως, αλλά δεν είναι απλή μια λύση όταν βρίσκεται κανεί στο χείλο τη χρεοκοπία. Σε πολλές λοιπόν χώρες κάποια στοιχεία των προγραμμάτων φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο απετυχημένα, αλλού πάλι κάποια στοιχεία ήταν επιτυχημένα. Σίγουρα δεν αντιμετωπίστηκε πλήρω η ανεργία ούτε οι κοινωνικέ επιπτώσει στι κοινωνίε των χωρών όπου υπήρξε λιτότητα, όμω κάποια ανάκτηση εμπιστοσύνη, κάποια επιστροφή των επενδύσεων, κάποια οικονομική ανάπτυξη ε, ήδη υπάρχει. Και σε κάποιε χώρε ήδη έχει να αντιμετωπίσετε και η ανεργία. Το αν είμαι πλήρω ικανοποιημένο, η απάντηση είναι όχι σε καμία περίπτωση όχι. Και αν πρέπει να επιτείνουμε τι προσπάθειέ μα σε όλου του τομεί τη ανάμειξη των πολιτικών μα, ναι, ναι, αλλά με τη σωστή ισορροπία και τη σωστή αναλογία. Η φύση τη κρίση που αντιμετωπίσαμε, που είχε πολλά να κάνει με τα και πληρωμών, και ε, τα εύκολα δάνεια, την ε, εύκολη διοχέτευση πιστώσεων στην προηγούμενη φάση είναι κάτι που για να αντιμετωπιστεί σε κρατικό επίπεδο θα χρειαστεί πολλή χρόνο. Δεν υπάρχουν λοιπόν μαγικέ λύσει και αυτό ε, θα πρέπει να το λέμε με ειλικρίνεια προ το κλικό μα σώμα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο πρώτο γύρο για τι πολιτικέ ομάδε και τώρα μπορούν να έχουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής αλλά έχουμε καθυστερήσει, έχουμε καθυστερήσει στο πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αλλαγή. Θα πρέπει να ε, έχουμε τις ερωτήσεις ανά τρεις, με ένα δίλεπτο για την κάθε ερώτηση και θα σας παρακαλέσω να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε και το πρόγραμμα. Ε, πρέπει να τελειώσουμε στις 10.30 γιατί ο κύριος Μπλουμ έχει και αλλού υποχρεώσεις πρέπει να ε, φύγει. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Θάλμπα Μπιντεγκάιν με τα κυρία Μπερέσ. Κύριε Πρόεδρε, τι έχουμε συνηθίσει εδώ, να υπάρχει αυστηρή πειθαρχία σε τέτοιε ακροάσεις από πάνω, από το Προεδρείο. Και θα το κάνατε. Και αν ε, συνεχίσουμε έτσι, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Θα πρέπει από την αρχή να εφαρμόζεται πιο πολύ πειθαρχία. Uh, ο Πρόεδρος. Δεν ε, είχαμε επιδείξει αρκετή πειταρχή, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι ο κατάλογος ομιλητός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές προκειμένου να πάρουμε και πιο πολύ χρόνο Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο όλη τη ομάδα Έκονα, αλλά το θέμα δεν είναι τα λίγα δευτερόλεπτα. Το θέμα ήταν ο κατάλογο ομιλητών που ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Α μην χάσουμε παραπάνω χρόνο, να δώσω πάρα αυτά το λόγο στον Παύλο Τσαλτομπελίκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Ντάζελμπλουμ που ήρθατε εδώ. Κύριε Ντάζελμπλουμ και μας δώσατε αυτές τις εξηγήσει. Η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι έφραυστη είπατε. Η ευθύνη μας είναι να αποφύγουμε αυτή η εύθραυστη οικονομία να οδηγήσει σε τελμάτωση. Επίσης, ε, μιλήσατε για τη σημασία ενός πώληση μίξ, ενός μείγματος πολιτικών. Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, είπατε ότι ελπίζετε να υπάρξουν περιθώρια λιγμού σε κάποιες χώρες, ώστε ε, να ακολουθήσουν ε, επεκτατικές, μια επεκτατική προσέγγιση. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις σημαντικές, θα ήθελα την άποψή σας για το κατά πόσον ε, λείπει η φιλοδοξία ε, από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους. Επίσης μιλήσατε για την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι δική της ευθύνη να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης και να προωθεί στην ανάπτυξη. Πράγματι μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο. Είναι αλήθεια όμως επίσης ότι και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, ο Μάριο Ντράγκη, δεν τρέφει και πολλές ελπίδες για το ότι θα αποδώσουν. Θα ήθελα επίση να μου πείτε αν εσείς ήσασταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα κάνατε κάτι παραπάνω από αυτά που κάνει μέχρι τώρα η ΕΚΤ. Τέλο, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Juncker, τι περιμένετε από αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο έχει ανακοινώσει ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κατευθυνθεί. Και σε ό,τι αφορά ε, το οχυρό αυτό, το ευρώ, αν αυτό επηρεάζει ε, το εύθραυστο της οικονομίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε του Eurogroup, ήδη σχολιάσατε την ομιλία του κύριου Ντράγκη Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει όμω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην ομιλία αυτή. Εδώ και καιρό μα εκκλείσει που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ασχολείται με το θέμα των μισθών. Και πλέον με την ομιλία αυτή και πέρα κάθε ενδεχόμενη ε, παρερμηνία, εδώ φαίνεται να ε, υπάρχει ουσιαστικά μία παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί μέσα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ενεργεία. Ε, ένα μεγάλο πρόβλημα τη Ευρωζώνη. Τώρα, στο φύλλο πορεία του κάθε κράτου μέλου ε, τίθενται κάποιε προποθέσει βάσει οικονομικών δεδομένων. Τα οικονομικά δεδομένα βάσει των οποίων όμω ε, προκύπτει και η εξέταση τη ανάπτυξη και η αναχώρα συστάσει είναι ε, πολύ σημαντικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου τη ετήσια δομή για τι προποθέσει του κάθε κράτου μέλου. Οι προποθέσει αυτέ λοιπόν έχουν αλλάξει πλέον. Θέλουμε να υπάρξει μεγάλη ε, μείωση του πληθωρισμού. Ε, βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη μείωση του πληθωρισμού ε, που δεν την είχαμε προβλέψει. Δεν ήμασταν καθόλου προετοιμασμένοι και οι προβλέψει ανάπτυξη δεν ήταν καθόλου στο ύψο των σημερινή κατάσταση που είναι πολύ χαμηλή η ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει έντονε προσπάθειε για διαρκωτικέ μεταρρυθμίσει που είναι πόδινε πολλέ φορέ. Αυτό θα ληφθεί υπόψη, ε, θα υπάρξουν στοιχεία ευελιξία που θα κινητοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι νέε συνθήκε, δείχνοντα ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε περπάνη. Και τώρα κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα σύντομο σχόλιο και ερωτήσει. Το σχόλιο μου έχει να κάνει με το ότι όταν βλέπουμε την τον αποπληθωρισμό, του κινδύνου των τελευταίων ετών. Βλέπουμε να μην είναι ένας κίνδυνο εθνικός ή κρατικός πλέον, αλλά ο κίνδυνος αποπληθωρισμού να αρχίζει να αφορά συνολικά την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι αν αντιμετωπίσουμε τον αποπληθωρισμό σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, δεν θα βρεθεί μια επαρκή λύση. Χρειάζεται μια συνολική απόκριση τη Ευρωζώνης μια μακροοικονομική πολιτική εδώ. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οικονομολόγοι που λένε ότι από αποπληθωρισμός και τα επίπεδά της στην Ευρωζώνη συνολικά θεωρείται ότι οφείλε, μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες. Δηλαδή και με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και με το Σύμφωνο ε, και Ανάπτυξης θα μπορούσε να υπάρχει ε, σύγκληση των ποσοστών εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Εσείς επίσης πώς αντιλαμβάνεστε την ε, ευελιξία και βάσει των ε, αντιδράσεων που έχετε από τα κράτη-μέλη. Επίσης για τη θεσμική διοργάνωση της Ευρωζώνης και σε σχέση με τις σημερινές μας προκλήσεις, τα σημερινά μας προβλήματα, ο συντονισμός των εθνικών αποκρίσεων στις αναχώρα συστάσεις. Κάτι που είναι δική σας ευθύνη, προσωπική ευθύνη και μια πρόκληση αρκε, αρκεί, αρκεί στο σημερινό πλαίσιο, στη σημερινή κατάσταση. Δεν χρειάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τέτοιες μακροοικονομικές πολιτικές. Μήπως θα πρέπει να υπήρχε μια νέα θεσμική διοργάνωση, ακόμα και από την πλευρά του Προέδρου της του Eurogroup, να υπήρχε πρόβλεψη θέσης ε, Προέδρου Ευρωζώνης λόγω χάρη. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε αυτές τις Ευχαριστώ κύριε Θάλμπα Πινταγκάνη για αυτές τις ερωτήσεις σας. Ναι, μπορεί κανείς να κάνει επικρίσεις εδώ, γιατί η προσέγγιση των ε, διαφόρων κρατών μελών στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεών τους είναι διαφορετική. Θα μπορούσαν κάποιοι να κάνουν περισσότερα. Οι χώρες βέβαια που ήταν σε μνημόνια σε πρόγραμμα λιτότητας έκαναν πολλά, άλλοι θα μπορούσαν να έχουν κάνει και περισσότερα. Λόγω χάρη η κυβέρνηση της Ιταλίας και της Γαλλίας, των νέες τους κυβερνήσεις, ήταν αρκετά φιλόδοξες στις μεταρρυθμίσεις τους, που μόλις όμως τώρα επιβεβαιώθηκαν από τις τα κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει περιθώριο αισιοδοξία. Όμως, κάποια από τα δρυφωτικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο 100 μελών. Λέτε, ο κύριος Ντράγκη δεν αφήνει περιθώριο ελπίδας. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα που έθιξε ο κύριο Ντράγκη είναι να μην τα περιμένετε όλα από την νομισματική πολιτική. Συμμορφωθείτε και κάντε ό,τι μπορείτε εντό του δημοσιονομικού σα περιθωρίου, χωρί να διαλύσετε το σύμφωνο προσέχοντα τα επίπεδα των επενδύσεών σα, ε, που μπορεί να είναι και δημόσιες εφόσον γίνεται, και ε, ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμό ε, τη δημοσιονομική συμπεριφορα στην Ευρώπη. Συμφωνώ με όλα όσα είπε, λίγο πολύ. Απλώ το βασικό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν λύσει και από την νομισματική πολιτική, αλλά και από την δημοσιονομική και ούτω καθεξή. Τώρα, για τα σχέδια επενδύσεων και αυτό που πρότεινε ο κ. Γιούνκερ, νομίζω η νέα Επιτροπή πολύ σύντομα θα έχει συγκεκριμένε προτάσει να υποβάλει, αλλά και εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν. Και εκεί λοιπόν θα καλυφθεί, θα καλυφθεί εν, μέρος, εν μέρη το πρόγραμμα, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα θεσμικά όργανα που ήδη διαθέτουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε εργαλεία και θεσμούς που ήδη υπάρχουν στη διάθεσή μας για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων. Για την κατάσταση του ευρώ Σίγουρα υπάρχει πτώση την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δύο εβδομάδες και η, μακρο... η βραχυπρόθεσμη και η μεσοπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά μα, οι προοπτικέ εξαγωγέ δεν επηρεάζονται άμεσα από αυτή την αλλαγή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή αποδυνάμωση που ίσω να είναι και διευκολυντική. Η ε, κυρία Περέσου. Μάλλον, είπατε μήπως ε, εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματικότητα. Νομίζω πως όχι. Πριν από 1,5 χρόνο υπήρχε αισιοδοξία για το πώς θα ανακτήσουμε το ρυθμό της ανάπτυξης. Τώρα, 1,5 χρόνο αργότερα, καταλαβαίνουμε ότι κάποιες από τις μεγαλύτερες χώρες έχουν κάποια σχετική παναχώρηση ω προς την μεγάλη αυτή ανάπτυξη που αναμέναμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα, η μεγάλη μας ανησυχία για όλους είναι μήπως παραμένουμε σε αυτό το τέλμα από οικονομικής σκοπιάς. Γι' αυτό πρέπει να αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως η ατζέντα των επενδύσεων που μόλις αναφέρα, η νομισματική πολιτική το πακέτο των μέτρων ε, για, τα, ε, για τους βασικούς φορείς από το Συμβούλιο πρέπει, τον Ιούνιο πρέπει ακόμη να υλοποιηθεί. Κάποιες χώρες βέβαια με την ευελιξία νομίζουν ότι αν ε, επικαλεστούν τον όρο αυτό θα λύσουν και όλες τα προβλήματα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Κυρία Χίμπνερ τώρα, μιλήσατε για τον κίνδυνο αποπληθωρισμού για την Ευρωζώνη συνολικά. Έχετε δίκιο έχει γίνει ένα πρόβλημα για την Ευρωζώνη συνολικά. Δεν βλέπω να υπάρχει κίνδυνος από πληθωρισμό ακριβώς, αλλά πολύ χαμηλός πληθωρισμός σε ένα μακρινότερο ορίζοντα. Αυτό πρέπει να κοπεί ως πορεία και εκεί νομίζω ότι υπάρχει κοινή ευθύνη για όλη την Ευρωζώνη για τις έκτακτες, ε, για τις εξαιρετικές συγκυρίες. Εδώ θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν τον Νοέμβριο συζητήσουμε τα σχέδια προπολογισμών. Εάν είναι πολύ χαμηλό ο πληθωρισμό και αν αυτό θεωρηθεί έκτακτε συνθήκε ω προ τα σύμφωνα, θα το δούμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη παρέκκληση από τι πρώτε εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ισχύσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν τα τωρινά επίπεδα χαμηλού πληθωρισμού μπορούν να σημάνουν κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει τη γνώμη της σχετικά. Και μετά θα τα συζητήσουμε και στο Eurogroup. Καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε κύριε Πρόεδρε της Ευρωομάδας. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας. Βέβαια δεν μπορώ να αξιολογήσω πολύ θετικά την ε, διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το εξής. Ουσιαστικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο γίνεται μια εθνική, ε, υπάρχει μια εθνική αντιμετώπιση και δεν λαμβάνονται υπόψη ε, τα αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα κάποιων εμπορικών πλεονασμάτων ορισμένων χωρών. Ε, μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα αυτό σε μια νομισματική ένωση γιατί επηρεάζει άμεσα τους εταίρους και πρέπει να το αξιολογήσουμε σωστά αυτό αλλά δεν υπάρχουν αυστηρές προειδοποιήσεις προς αυτές τις χώρες. Με αυτή την προσέγγιση έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα. Ε, το εξάμεινο αυτό δεν έχει μία ανάλυση του πώς προχωρά η νομισματική ένωση και δεν γίνεται συζήτηση για τις πραγματικές διαθροτικές μεταρρυθμίσεις ευρωζώνης. Πρέπει να έχουμε μία δημοσιονομική πολιτική σωστή να προχωρήσει η ενιαία αγορά αλλά ε, θέλουμε μια καθολική προσέγγιση μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει μια μεταφορά εξουσίας από τις χώρες προς την Ένωση με σημαντικό κοινοβουλευτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η μεταφορά εξουσίας είναι η μόνη λύση για να υπάρξει ε, η λαϊκή κυριαρχία εκ νέου. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν σε επίπεδο κρατών. Αυτή είναι η γενική μου προσέγγιση. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να λυθεί η κρίση μόνο με εθνικές μεταρρυθμίσεις από τις χρωμένες οικονομίες, η νομισματική πολιτική και επεκτατική βέβαια αν γίνει, θα αρκέσει για να λυθούν τα προβλήματα θα υπάρξει αύξηση, θα υπάρξει ανάπτυξη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή δημοσιονομική αναπτυξιακή πολιτική και δημοσιονομική δέσμευση από τις χώρες που έχουν μεγαλύτερα περιθώρια λιγμών. Και τέλος, ένα γραφειοκρατικό ερώτημα. Θεωρείτε ότι η Προεδρία του Eurogroup θα πρέπει να είναι ένα πλήρες κατά κάποιο τρόπο αξίωμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέρνερ Κύριε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας κάνω ένα κομπλιμέντο για το πώς έχετε προασπίσει τις αποφάσεις σας την τελευταία ώρα εδώ. Πραγματικά εκπληκτικό. Τρεις μικρές ε, ερωτήσεις. Ε, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί περαιτέρω η νομισματική πολιτική. Μπορείτε να λέτε ότι θέλετε ανεξαρτησία των Ευρωπαϊκών Κεντρικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά ο κύριος Ντράγκη δεν είπε τίποτα καινούριο. Εκφράστηκε για το πρόγραμμα του Juncker, για το συντονισμό της Ευρωζώνης για τι υιοθετικέ μεταρρυθμίσει των κρατών. Δεν είπε τίποτα το καινούριο, αλλά υπάρχει η κίνηση στις ε, άλλου τομείς ε, ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό ε, διαφορετική κατεύθυνση η νομισματική πολιτική. Η Λιθουανία θα γίνει το 19ο κράτος της Ευρωζώνης και θα έχουμε 7 χώρε με ε, ρυθμίσεις έκτακτες. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι θα διαμορφωθεί και η περαιτέρω προσχώρηση στην Ευρωζώνη και τρίτον για τον φορολογικό συντονισμό. Ως πρόεδρος της Ευρωζώνης και ως ε, ε, Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας σας ε, ρώτησαν για το Irish Dutch Package για την νόμιμη αποφυγή, φοροαπηφυγή όπου οι σχετικές άδειες δεν φορολογούνται ή φορολογούνται πολύ χαμηλότερα και έτσι οι 10 μεγαλύτεροι οργανισμοί του διαδικτύου έχουν ε, έδρα στην Ιρλανδία, έξω από το Διβλίνο και παίρνουν άδειε στην Ολλανδία. Προτίθεστε να τα σκεφτείτε αυτά τα θέματα και πώς θα, αντιμετωπίσετε, πώς θα αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάισελμπλουμ, έγινε πολύ λόγο για τι ιδιωτικέ και δημόσιε επενδύσει για την Ευρώπη και όλοι λένε ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο να έχει μακροπροθέσιμου στόχου. Η δική μου ερώτηση είναι να μου πείτε την άποψή σα για ένα τεχνικό πρόβλημα για τι μεγάλε επενδύσει διότι για μένα ο νέος κανόνας αναφοράς για την ανάλυση και το αν θα λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες επενδύσεις δεν, ε, αφήνει να, δεν κάνει σαφές το αν θα είναι σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σωστός υπολογισμός στο χρέος των επενδύσεων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπει κανείς τι γίνεται και με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Στη χώρα μου το Βέλγιο 50% των δαπανών ως επενδύσεις μπορεί να οδηγούν σε ελάχιστο 5% από το κρατικό χρέος στον υπολογισμό. Το 2000-2014 όμως όχι απλώς δεν ενθαρρύνθηκαν οι ε, ε, κυβερνήσεις αλλά ουσιαστικά υποχρεώθηκαν έτσι εξαρτάται άμεσα το ποσοστό του χρέους από το πώς ε, γίνονται επενδύσεις. Δηλαδή καλύπτεται ένα τρέχον έλλειμμα από τις επενδύσεις που γίνονται, αντί να εξυπηρετεί σωστή στόχη. Γι' αυτό η αξιολόγηση όπως γίνεται με οικονομικούς όρους δεν είναι η σωστή και δεν φαίνεται αν υπάρχει χρηστή διαχείριση ή όχι από ένα δημόσιο φορέα. Ένα παράδειγμα, χάρη στα Ευρωπαϊκά Διαπρακτικά Ταμεία, λόγω χάρη στην κοινότητα μου, δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε ένα ε, πάρκο στην περιοχή, αλλά δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει την ε, ε, επένδυση αυτή για να φτάσει στο τέλος του το έργο, διότι θα φτάσει στο μέγιστο επίπεδο χρέωσης. Θεωρείται λοιπόν ότι θα μπορούσαν να είναι οι δημόσιες επενδύσεις ενεργητικό και να μην υπολογίζονται πλέον στο χρέος. Και Πώς θα υπολογίζονται οι επενδύσεις εφόσον θέλουμε να υπάρχει οικονομική ανάκαμψη και διάσωση και να μην ε, περιλαμβάνονται στους κανόνες για το Μουσουλμικό Συμφώνο. Και επειδή όλοι μιλήσαμε για το λόγο του κ. Ντράγκη, είπε ότι πρέπει να ε, συμμορφώνεται κανείς όχι μόνο με τους κανόνες του Δημοσιονομικού Συμφώνου, αλλά ότι χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο δημόσιων επενδύσεων. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και πώς θα υλοποιηθεί εάν τις δαπάνες για τις επενδύσεις, τις δημόσιες επενδύσεις δεν τις λάβουμε και δεν τις υπολογίσουμε σωστά. Πρόεδρε. Thanks Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φερνάντες Αλβάρε, μιλήσατε για μια κατάσταση όπου μόνο οι εθνικέ μεταρρυθμίσεις θα μα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Η απάντηση είναι όχι. Όχι, δεν θα είναι μόνο οι εθνικέ ε, ε, μεταρρυθμίσεις, όπω δεν μπορεί να είναι μόνο η νομισματική πολιτική αυτή που θα μα οδηγήσει στη λύση. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει στην ερώτηση του κ. Λάγκα για την νομισματική πολιτική. Νομίζω ότι ήδη έχουμε οδηγήσει σε νέες κατευθύνσεις στη νομισματική πολιτική, απλώνοντας τις δυνατότητες με τρόπο καινούριο. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον Εμένα Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Σε καινούργιες λοιπόν κατευθύνσεις έχουμε διοχετεύσει την νομισματική πολιτική. Αλλά εδώ θα συμφωνήσω με τον Μάριο Ντράγκη ότι δεν είναι δυνατόν η λύση να έρθει μόνο από την νομισματική πολιτική. Αυτό θα ενήχει κάποιου κινδύνου, του οποίου δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε. Και πάλι, θέλουμε μείγμα μεταξύ εθνικών ε, ευθυνών, εθνικών ε, μεταρρυθμίσεων, συντονισμού μεταρρυθμίσεων για όλε τι χώρε στην Ευρωζώνη και αυτά τα αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Ευρωζώνη, Eurogroup υγιούς πολιτικής ε, χρηματοοικονομικής που θα περιλαμβάνει και ευελιξία μέσα στα δεδομένα όρια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν το στόχο μας με τη νέα Επιτροπή και η νέα Επιτροπή έχει εκφράσει την προθυμία και την διάθεση να προωθήσει σχέδια επενδύσεων. Τελευταία ερώτηση. Κατά πόσον θα πρέπει να αποτελεί αυτό κάτι το μόνιμο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και είμαι πολύ ανεκτός σε ό,τι αφορά θέματα διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Αλλά πρώτα το θέμα θα πρέπει να είναι το τι είδους φιλοδοξία θέλουμε να επιφέρουμε και πόσο μακριά θέλουμε να πάμε, σε τι βαθμό θέλουμε να μεταφέρουμε αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες, σε ποιους τομείς και ε, ένα στοιχείο αυτών των συζητήσεων στη τελική ανάλυση θα πρέπει να είναι πού θέλουμε να καταλήξουμε με τις ε, θεσμικές μας, τα θεσμικά μας όργανα. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη αντιπροσωπεία με, μόνιμο, με μόνιμους υπαλλήλους, μόνιμο πρόεδρο. αλλά δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητες και τι ευθύνε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Α γίνει όμω αυτή η συζήτηση για το πολιτικό περιεχόμενο. Α γίνει αυτή η συζήτηση για τι πολιτικέ ευθύνε προτού οικοδομηθούν νέοι θεσμοί. είναι, αυτή είναι η σωστή ο, σειρά. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Λάγκε. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική, ήδη επιτυκνύουμε αρκετή καινοτομία σε ό,τι αφορά τη μελλοντική προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Όπως θα ξέρετε, ήδη έχουν προσχωρήσει καινούργια μέλη σε μία περίοδο όπου μιλούσαμε για κρίση της Ευρωζώνης και αυτές οι χώρες απέδειξαν ότι είναι πολύ αποφασισμένες και ότι θεωρούν την Ευρωζώνη τμήμα της σταθερότητάς τους, της πολιτικής σταθερότητάς τους, της οικονομικής τους σταθερότητάς και υποστηρίζουν τις χώρες της Βαλτικής στην πεποίθησή τους ότι σε ό,τι αφορά την μελλοντική του σταθερότητα, πολιτικός και οικονομικός πώς, το να ανήκουν στην Ευρωζώνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας και εγώ αναμένω αύξηση, διεύρυνση της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θα το καλωσόριζα. Για την νόμιμη φοροαποφυγή. Αγαπημένο θέμα. Με χαρά μου σας λέω ότι η Ολλανδική κυβέρνηση έχει λάβει κάποια μέτρα για τα στοιχεία που αναφέρεται, Για παράδειγμα, γιατί τόσε διεθνεί επιχειρήσεις έρχονται στη χώρα μας, γιατί έχουμε μεγάλο όγκο φορολογικών συμφωνιών. Και τώρα τις αλλάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αφαιρεθεί το στοιχείο της δυνατότητας της φοροαποφυγής, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η δυνατότητα. Αλλάζουμε λοιπόν μεγάλο τμήμα των ε, συμφωνιών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι σοβαρό και το αντιμετωπίζουμε. Τέλος. Κύριε Μπάγετ. είπατε ότι οι τοπικέ κυβερνήσει θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν. Νομίζω ότι το κάνουν. Αλλά θεωρώ ότι ρεαλιστικά θα πρέπει να δούμε ότι τα επίπεδα χρέωση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται το επίπεδο χρέωσης μια ολόκληρης χώρας, γιατί αυτό μακροπρόθεσμα είναι μεγάλος κίνδυνος για την ε, σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Ντάισελμπλουμ στην Επιτροπή μας, η οποία είναι καινούργια Επιτροπή για μένα, αλλά έχουμε συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό ω πρόεδρο τη Ευρωζώνη. Του εύχομαι ό,τι καλύτερα για την υπόλοιπη θητεία του και για τη μετέπειτα φάση. Θα ήθελα να πω ότι στον πρόεδρο. Στο τέλος είπατε ότι οι εξαιρετικές θυσίες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και στη δική μου και στην Πορτογαλία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και τώρα χώρες όπως η Πορτογαλία έχουν επανέλθει στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι σημαντικό να παραμείνουν. Μία από τις προτάσεις η οποία έχει κατατεθεί προσφάτως είναι ότι σε ό,τι αφορά το τμήμα και το σκέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της ε, Τρόικας, οι χώρες όπως η Ιρλανδία θα μπορούσαν να ξεπληρώσουν ε, εγκαίρως, πρόημα, το χρέο του προ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά τίθεται και θέμα αρεσιμότητα, Να σα ρωτήσω ποια είναι η γενική σα θέση για την άποψη αυτή. Δεν θα έχει νόημα χώρε οι οποίε ήταν σε μνημόνια και θέλουν να πληρώσουν, να τα αποπληρώσουν πιο νωρίς με χαμηλότερο επιτόκιο να μπορούν να το κάνουν και πώς η Ευρωζώνη, το Eurogroup πρόκειται να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Τάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε Πρόεδρε του Eurogroup. Πρώτη φορά βρίσκεστε εδώ μετά τι εκλογέ. Οι εκλογέ στην Ολλανδία ε, αφορούσαν πολύ τα χρηματοπιστωτικού ε, κανόνε. Η χώρα μα ε, και το κόμμα μα πρότεινε να μην υπάρχει μόνο κανόνα για το έλλειμμα αλλά και για την ανεργία γιατί αναζητούμε τρόπου να έχουμε αξιόπιστη χρηματοπιστωτική πολιτική αλλά και ευελιξία την ίδια λοιπόν ε, προσέγγιση που ακολουθείται στο διάλογο αυτό. Να επανέλθουμε σε μία από τις αντιπαραθέσεις με τον ίδιο Μπούλμαν. Πώς θα συνδυαστεί η αξιοπιστία με την ευελιξία σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις ε, δημόσιες επενδύσεις ε, που θα μπορούσαν ενδεχομένω να έχουν πιο πολύ χρόνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρηματοπιστωτικό έλλειμμα. Σας παρακαλώ, για να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, υπάρχετε. θέλετε να υπάρξει μια επίσημη ε, ε, διαδικασία, θέλετε να αναλάβετε μια πρωτοβουλία για να υπάρξει αυτή η εγγύηση ευελιξίας και ε, τήρησης των κανόνων. Ευχαριστώ, Μορεζάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάισελμπλουμ, καλώ ήλθατε στην Επιτροπή μα. Σα καλωσορίζουμε. Και εμεί, βέβαια, ω νέα μέλη, για πρώτη φορά μπορούμε να ανταλλάξουμε μαζί σα απόψει και είμαστε ευγνώμονε γι' αυτό. Είπατε ότι η απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να προέλθει μόνο από την ΕΚΤ, αλλά χρειάζεται ένα ευρύτερο μείγμα πολιτικών και βέβαια συμφωνώ μαζί σα. Επίση, πολύ σωστά είπατε ότι η ΕΚΤ από μόνη τη θα αποφασίσει εφόσον και πού θα κάνει παραπάνω θα, θα λάβει περισσότερα μέτρα. Σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, ε, το ερώτημά μου και την ενδεχόμενη παρέμβαση της ΕΚΤ, το να κάνει περισσότερα στο πλαίσιο που παραδείγματος μιας ποσοτικής χαλάρωσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα ε, δάνεια από τις τράπεζες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, σε μεγαλύτερη κατανάλωση από τους πολίτες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι προϋπόθεση για μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μια τέτοια παρέμβαση θεωρείτε ότι θα μειώσει ε, τα κίνητρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όχι. Και τελευταίο ερώτημα, αν αποφασίσει να παρέμβει ΕΚΤ, βλέπετε κίνδυνο μιας φούσκας ε, στις τιμές ε, του ενεργητικού. Να απαντήσετε κύριε Με Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Χέις. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημαντική σας νέα θέση. Το ερώτημά σα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αφορούσε τα δάνεια του Νιτάφ για την Ιρλανδία. Ξέρουμε ότι εξετάζουν ενδεχόμενο πρόορις αποπληρωμής αυτών των δανείων. Και αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλο όφελο σε ό,τι αφορά ε, τους στόχους που δεν θα καταβάλει Είχα μια επαφή με τον Ιρλανδό Υπουργό και με άλλους θεσμούς, με άλλους φορείς. Μου είπαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτό. Νομίζω θα το συζητήσουμε το Σεπτέμβριο, την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, σύντομα δηλαδή θα το, θα το δούμε με βάση αυτό το αίτημα της Ιρλανδίας, που επισήμως δεν έχει κατατεθεί ακόμη, γι' αυτό και πολύ προσεκτικά διατυπώνω την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αιτηθούν επισήμως το ε, μέτρο και μετά θα συζητηθεί από το ΕΚΟΦΗΝ και θα πρέπει να εγκριθεί αυτό το αίτημα. Για να ξεκινήσει το η πρόορη αποπληρωμή μόνο του σκέλους ε, του δανείου του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Αυτό που σας ενδιαφέρει λοιπόν, ναι, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ιταλία, στη συνεδρίαση του Eurogroup. Τον κύριο Τάγκ, που τον γνώριζω πολύ καλά γιατί ήμασταν ε, βουλευτέ ε, στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και οι δύο. Μου είπατε να μιλήσω πιο πολύ για την ευελιξία σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Ακούστε, στο πλαίσιο του συμφώνου φυσικά Έχουμε το διορθωτικό και το προληπτικό σκέλος και κάνουμε διάκριση μεταξύ των δύο. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για το τι σημαίνει ευελιξία στα δύο αυτά σκέλη. Στο διορθωτικό σκέλος υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων κτλ. κτλ να δοθεί μεγαλύτερος χρόνος στις χώρες για να πετύχουν τους στόχους. Δικό μου αίτημα θα ήταν, εάν δοθεί έξτρα χρόνο, βάσει των όρων και προποθέσεων που προανέφερε, να μην χαθεί ο χρόνο αυτό, αλλά να αξιοποιηθεί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ε, χώρα, την εκάστοτε να ορίσει τις μεταρρυθμίσει, οι οποίε θα πρέπει εμπροστοβαρός, αν θέλετε, να, εκ των προτέρων δηλαδή, να μπουν στη μέση διάταξη. Στο προληπτικό σκέλος, από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα πιο πολύπλοκο δίκτυ για το διαρθωτικό έλλειμμα. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 6-pack και του 2-pack, εξάπτυχου δίπτυχου. Έχουμε τον ενδιάμεσο στόχο μας βέβαια, άρα μπαίνει και εκεί το στοιχείο του χρόνου, ενδιάμεσος στόχος, μεσοπρόθεσμος στόχος. Κάποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν και να, να φαίνονται και στον προπολογισμό. Χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη αυτό το στοιχείο του χρόνου στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων όταν θα υπολογίσουμε τον, τον μέσο πρόθεσμο στόχο για μια χώρα. Βάσει δηλαδή των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την λόγο χώρα θα αποφασίσουμε και τον μέσο πρόθεσμο αυτό στόχο. Αλλά έκανα τη σαφή διάκριση μεταξύ του διορθωτικού σκέλους αφενός και του προληπτικού σκέλους αφετέρου. Και ελπίζω όλο και περισσότερες ε, χώρες να στραφούν στο προληπτικό σκέλος, ώστε αυτή η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο στόχο και τις μεταρρυθμίσεις να γίνεται όλο και πιο σημαντική και αυτό να μας απασχολεί περισσότερο. Αυτά έχω να πω σε αυτό το θέμα. Τέλος, προς τον κύριο Μιρεσόνη κάπως έτσι, είπατε ότι χαίρεστε που είπα ότι δεν θα δοθεί απάντηση μόνο από την ΕΚΤ. Και τονίζω το μόνο. Γιατί ρόλο σημαντικό έχει να διαδραματίσει και τον διαδραματίζει. Επίση, είπατε ποιε μπορεί να είναι οι συνέπειε περισσότερη ποσοτική χαλάρωση. Πρώτα απ' όλα, λάβουμε κάποιε αποφάσει τον Ιούνιο. Αυτέ οι αποφάσει πρέπει να υλοποιηθούν. Και αυτό θα γίνει μέσω των διάβλων χρηματοδότηση. Δεν έχει γίνει ακόμη. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα της μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Κίνδυνος, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει. Εάν βγάλουμε έξω πολύ φθηνό χρήμα, κίνδυνος να δημιουργηθούν φούσκες στην πραγματική οικονομία. Και έτσι να αποβεί αυτό σε βάρος της οικονομίας μακροπρόθεσμα, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ λογικοί και προσεκτικοί με αυτά που κάνουν. Να μην βασιστούμε πάρα πολύ στην νομισματική πολιτική, γιατί εκεί ε, ενέχουν, ελοχεύουν κίνδυνοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γερούν, σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι επιτελέσαμε πρόοδο, καταλάβαμε κάπως καλύτερα και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας για την ευελιξία. Επόμενη συνεδρίαση στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Θα σας δω λοιπόν σε δύο εβδομάδες. Λίγη συνεδρίαση.